Good morning everyone. Καλημέρα σε όλους σας. Σας παρακαλώ να καθίσετε και να ετοιμάσετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας, γιατί θα αρχίσουμε με ψηφοφορίες μεμονωμένες, τις οποίες και θα διεξαγάγουμε ηλεκτρονικώς. Okay, so the first vote. Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία. On uh, the provisional agreement. Για την προσωρινή συμφωνία. Spirit drinks. Για τα πνευματόδη. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας και πάλι. Αυτή τη φορά αφορά τις εκπομπές ε, διεξουδίου του άνθρακα ε, από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αρχής ψηφοφορία και τα ταχύ Πέρας. Εγκρίνεται. Now we vote on the provisional agreement. Τώρα ψηφίζουμε την προσωρινή συμφωνία για τα πλαστικά μια χρήσεως. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Now we are uh, voting on a draft motion. Τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος για διάφορες αντιρρήσεις που έχουμε για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. And it's closed. εγκρίνεται. This, the same thing, this time... Η ίδια ψηφοφορία για τον αραβόση του τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Again, Επόμενη ψηφοφορία, πάλι ένα ψήφισμα για τον τροποποιημένο ή το μόνο 87403, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία για το γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι. Αρχίζει ψηφοφορία. Τώρα θα ψηφίσουμε μια προφορική ερώτηση σχετικά με τη στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. That says commission again. That's okay. Now we are voting on the... Τώρα την ίδια προφορική ερώτηση θα ψηφίσουμε, αλλά προς το Συμβούλιο αυτή τη φορά. Αρχίζει η ψηφοφορία. And it's closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Now we are voting on a draft opinion. Τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινή δήλωση που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές η CR είναι υπέρ εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος της 30 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 31 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, έλεγχος του πρώτου τμήματος. Αρχίζει τώρα, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ. Against. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά θα αρχίσει τώρα. Closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Now we are voting on a draft. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις ε, και προϋποθέσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Wow. Λοιπόν, μητροπολογία 114 ψήφι υπέ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 1 υπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 229 υπέρ κατά έλεγχο σας παρακαλώ. Πέρας. Rejected. Απορρίπτεται. 2.23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.37 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 29 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχο σας παρακαλώ. Πέρας εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει 261 και προχωρούμε στη 277 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Παρακαλώ. 2,77. Πέρας. Απορρίπτεται. 78 in favor. 2,78 υπέρ. Against abstentions adopt. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2,83 και άγκρι 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2,92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 40 υπέρ Against. Abstentions adopt. κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει συμβιβαστική 5α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπράβο σας κυρία Μποναφέ, πολλές συμβαστικές έχετε. 3.39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3.40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 341 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 353, όχι, έχουμε τη συμβαστική 14 προηγουμένως. Ψηφί υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 353 υπέρ, κατά. Το ΕΛΚ τι λέει, υπέρ είσαστε ή κατά. Υπέρ, ωραία, τότε εγκρίνεται. Η 46 ε, της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές. Και πάλι δεν βλέπω τι λέει το ΕΛΚ. Υπέρ είστε, ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 54 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 391 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 395 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 396 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 398 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 400 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η άγκρη 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 401 όχι έχει καταπέσει, 404 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Η συμβαστική 10 υπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 408 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 409 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 410 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 411 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η άγκρι 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 66 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 67, όχι δεν την ψηφίζουμε. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 426 in favor. 426 υπέρ, κατά. Το ΕΛΚ τι ψηφίζει. Εγκρίνεται ωραία. 30, who in favor. 430 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 431 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 434 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 438 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 88 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ. The vote is closed. Adopted. 439 υπέρ. Ε, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 440 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 441. Μη προσθήκη. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 443 υπέρ. No, this falls. 444. πίπτη, συγγνώμη. 444 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Against. Κατά αποχές εγκρίνεται. 446 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 447 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Agri one, who is in favor. Η ένα της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 in 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά το ΕΛΚ τι ψηφίζει υπέρ κρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 ψηφί υπέρ κατά αποχές. Επανάληψη παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 4-4, 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές. Η πράσινη, η γκουε, η καναχέρι. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Η τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 17 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πού είμαστε τώρα? 175. σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ, εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ, κατά έλεγχος. The Πέρας και απορρίπτεται. 18 Η Άγκρη 18 έχει μια προφορική τροπολογία την οποία βλέπετε εδώ γραμμένη. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς με αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Άρα θα τεθεί σε ψηφοφορία. Δηλαδή ψηφίζουμε τη 18 μαζί με την προφορική τροπολογία. Ψήφι της τροπολογίας 18 της Επιτροπής Γεωργίας με την προσθήκη της προφορικής τροπολογίας. Κατά αποχές εγκρίνεται. 179 ΕΠΕ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 ΕΠΕ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 ΕΠΕ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 ΕΠΕ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 21 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 και άγκρι 23 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 198 ψηφίζουμε, μάλιστα 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται «201 υπέρ,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 κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 και άγκρι 26 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική αρχίζει τώρα. And it is closed. Εγκρίθηκε Now we are voting on a draft report on implementation. Θα ψηφίσουμε ε, το σχέδιο έκθεσης για την εφαρμογή ε, της οδηγίας ε, για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Amendment 70. 70. Ποιος είναι υπέρ? Κανείς. Κατά. Απορρίπτεται. Ήμκο 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 2 υπέρ όχι, όχι συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ α όχι έχει αποσυρθεί συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά ηλεκτρονική επιβεβαίωση. The vote is closed.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 EPP is against. Check. The vote is over. εξακριβωση εξακρίβωση. Cross-party association. It is... Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά εποχέ. εγκρίνεται. Ήμκο α υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ήμκο d υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ήμκο e υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά εποχέ, εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 3 ε, συμβαστική 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 22. 2 υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Όχι. Όχι, όχι. Δεν επιμένω. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. And it's closed. υιοθετείται η έκθεση. Πολλές ε, συμβαστικές τροπολογίες. Περνάμε την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2009-128 για σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωρικών φαρμάκων. Ξεκινάμε με την τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Άγκρι 2 υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. εγκρίνεται εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά εποχές ε, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά εποχές απορρίπτεται. Ε, εξακρίβωση, ηλεκτρονική εξακρίβωση. Ίσως οι φιλελεύθεροι να με παραπλάνησαν. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία άγκρη 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Υπέρ. Κατά αποχές Ας το ας κάνουμε ηλεκτρονική εξακρίβωση. Λήξη πληροφορία εγκρίνεται 90. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά ελεύθερη, φιλελεύθερη κατά απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές Ελεκτρονική εξακρίβωση λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. ...146 υπέρ... ...κατά... ...αποχές εγκρίνεται... ...147 υπέρ... ...κατά... ...αποχές απορρίπτεται... ...148 υπέρ κατά εποχές έλεγχος ηλεκτρονικός έλεγχος And it is uh, closed. Λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. εποχέ, απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Το ΕΛΚ τι είναι υπέρ κατά. Οπότε εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Άγκρι όχι. 167 υπέρ. Κατά, Εποχέ. απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά, Εποχέ. απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά, Εποχέ. απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά, Εποχέ. απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά, εποχέ απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά, Εποχέ. απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ κατά πράσινη υπέρ κατά είστε. 194 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Άρχιτη η ψηφοφορία. It's closed. Εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Mr. Housing is not happy. It's closed. It's closed. Λήξη ψηφοφορία εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. Άγκρι 18 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά εποχέ απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 2.25 υπέρ κατά εποχέ, εγκρίνεται 2.23 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.37 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.38 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 2.41 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.50 και 2.51 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 2.52 υπέρ. Κατά. εποχές, απορρίπτεται. 2.53 υπέρ. Κατά. εποχές, απορρίπτεται. 2.54 υπέρ. Κατά. εποχές, απορρίπτεται. 2.55 υπέρ. Κατά. εποχές, απορρίπτεται. 2.56 υπέρ. Κατά. εποχές, απορρίπτεται. 2.57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.58 και άγκρι 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.60 υπέρ κατά εποχέ, εγκρίνεται. Άγκρι 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.62 υπέρ κατά εποχέ, εξακρίβωση. Άρχεται.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 εγκρίνονται. 5 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται ή όχι. Εγκρίνεται. 6 και 7 μαζί υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 8 και 9 μαζί υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, τη 12. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται 23 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται 24 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται 25 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται 26 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται Εγκρίνεται. Okay, now we are going to vote on... Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο νομοδοτήσεων για τις απαλλαγές. <laughs> um, the first one is on European... Η πρώτη αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είστε έτοιμοι να οματοποιήσουμε τις ψηφοφορίες για τις απαλλαγές. Εν πάση περίπτωση, η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ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 η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Άλλη απαλλαγή. Εύσα. Οργανισμός τροφίμων. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές. Οι φιλελεύθεροι τι κάνουν. Υπέρ είναι κατά. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 σε 2 τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 5 σε 2 τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 υπέρ, κατά, απόχες η άλλη είναι αντίθετη ή υπέρ. Δεν έχω καταλάβει. Αφήστε τους να απαντήσουν ε, οι πράσινοι εμέσως. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 7. Ε, υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 8. Α, την 6 θέλετε να τσακάρουμε. Ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 6. Πέρας. Είπατε είστε κατά. Έτσι, εγκρίνεται. Η τροπολογία 9 τώρα. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά τώρα αρχίζει και τελειώνει και εγκρίνεται. Προχωρούμε. Απαλλαγή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Έχουμε τρεις ψηφοφορίες εδώ, τις απολογίες 1, 2, 3 μαζί, Είπε κατά, αποχές, απορρίπτονται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα και τελειώνει αμέσω και εγκρίνεται. Άλλη απαλλαγή για την ε, έχα των χημικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, πέντε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία αρχίζει τώρα και λίγη και εγκρίνεται η απαλλαγή. Η έκθεση. Η ΕΜΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες μαζί. 1, 2, 3, 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Και τελειώνει κιόλας και εγκρίνεται. Άλλη απαλλαγή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Τέσσερις ψηφοφορίες ομαδοποιημένες και αυτές. Τροπολογία 1, 2, 3, 4. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Και τελειώνει επίσης και εγκρίνεται η έκθεση και τελειώσαμε πριν τις 11, τα κατάφερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. At 11.15 we have uh, the minister. και έρχεται ο υπουργο Γεωργίας της Ρουμανίας, ή Υπουργό, συγγνώμη. Έχετε παρακαλώ ε, διάλειμμα ένα τέταρτάκι. Συγγνώμη, ο υπουργο Γεωργίας. Let's uh, start our Μπορούμε να ξαναρχίσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας που κατέχει την Προεδρία Εκπεριτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. Έχουμε. εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να συζητήσουμε θέματα της κοινή μας ατζέντα περιβάλλοντος και γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να μας κάνετε μια παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας σε αυτό το τομέα. Αγαπητή Αντίνα, ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισήγησή σας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μία αγαστή συνεργασία και θα ήθελα να σας κάνω μία παρουσίαση των προτεραιοτήτων μας. Είναι μεγάλη τιμή μου. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι μεταξύ σας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας. Θα ήθελα να απευθύνω τον χαιρετισμό του αγροτικού κόσμου της Ρουμανίας, της βιομηχανίας τροφίμων και των καταναλωτών που ευεργετούνται από τις ε, πολιτικές σας. Για την Ρουμανική Προεδρία αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πρώτη φορά ασκούμε την Προεδρία 12 χρόνια μετά την προσχώρησή μας. Πρόκειται για μια δυναμική πορεία με μία σειρά γεγονότων που θα έχουν μία αλληλουχία και ελπίζω να μπορέσουμε να είμαστε ένας αμερόληπτος διαμεσολαβητής. Η διάσκεψη στο Συμπίου της 9ης Μαΐου 19 θα αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο για να είμαστε πιο ενωμένοι και πιο συνεκτικοί και δημοκρατικοί. Αυτό το γεγονός θα βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που είναι απόλυτα αναγκαίες για την παγιοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος. Θα ήθελα να κοινοποιηθεί καλύτερα η ευρωπαϊκή ατζέντα στους πολίτες. Η Ρουμανία θα προωθήσει αυτά τα σχέδια σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να ευεργετηθούν όλοι από μία δυνατή ένωση η οποία να είναι συνεκτική και αποδοτική. Επίσης, η Ρουμανική Προεδρία θα παρακολουθήσει και θα ακολουθήσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της συνοχής και των περιφερειών. Πιστεύουμε ότι η συνοχή είναι μια κοινή αξία που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Την Ευρώπη της σύγκλησης, την Ευρώπη της ασφάλειας, της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα και της Ευρώπης των κοινών στον πρώτο πυλώνα στην Ευρώπη της Συνοχής θέλουμε να προωθήσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη για όλους τους πολίτες με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την μείωση των ανισοτήτων, την προώθηση της ψηφιοποίησης και του επιχειρήν. Στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα όσον αφορά την Ευρώπη της ασφάλειας, θέλουμε να έχουμε μια πιο ασφαλή Ευρώπη έναντι των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφαλείας και των απειλών. Σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα, ο γενικός στόχος είναι Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγων να προωθήσει την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής με τους κατάλληλους, κατάλληλους πόρους για να προωθήσουμε και τις δράσεις της Ένωσης στην πολιτική γειτονίας. Σε σχέση με τον τέταρτο πυλώνα, ο γενικός στόχος αφορά την προώθηση της αλληλεγγύης και της συνοχής μέσω πολιτικών για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, των διακρίσεων και για τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και την προώθηση του γίγνεσθε για να ευεργετηθούν οι πολίτες. Αυτά μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 θέλουμε μέσω προϋπολογισμού να φτάσουμε στους στόχους κατά την επόμενη επταετία. Οι δεσμεύσει της Προεδρίας σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο προωθούν τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί πρόκριμα για τα τελικά αποτελέσματα. Θα θέλαμε επίσης να προωθήσουμε την συνοχή μεταξύ όλων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ευρέως γνωστή, εκπροσωπεί τους πολίτες, κάτι το γνωρίζω πολύ καλά και υπό το προσωπικό πρίσμα, διότι ήμουν ε, μέλος της ε, Επιτροπής Γεωργίας στο Εθνικό Κοινοβούλιο για 12 χρόνια και πρόεδρος της Επιτροπής για 4 χρόνια. Σας εγγυώμαι λοιπόν ότι είμαι διαθέσιμος για να συνεργαστώ μαζί σας επικοδομητικά και αποτελεσματικά για να προωθήσουμε τα ε, διάφορα νομοθετικά σχέδια σε επίπεδο ένωσης και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελίσαπεθ Κέστιγκερ για τη συνεργασία και γιατί κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα επίσης να σε συγχαρώ αγαπητή Αντίνα μαζί με ολόκληρη την ομάδα σου για την διενέργεια διαπραγματεύσεων και μέσα στα πλαίσια των εκρεμών υποθέσεων νομοθετικού περιεχομένου. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές, γνωρίζοντας ότι διαθέτουμε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να φτάσουμε σε μία συμφωνία και για να ολοκληρώσουμε μέσα σε αυτή τη θητεία τα κείμενα νομοθετικού περιεχομένου. Ο χρόνος ε, είναι ο μεγάλος μας εχθρός. Είμαι πεπισμένος όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Βασίζομαι στην αγαστή συνεργασία στα πλαίσια του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, θα πρέπει να είναι οι μεγάλοι εμπλεκόμενοι αυτής της διαδικασίας. Και αυτό αφορά και την ε, ασφάλεια τροφίμων, την προστασία της ανθρώπινης υγείας, των ζώων και του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα τρόφιμα να είναι ποιοτικά, να εξασφαλίζουν τις ε, βασικές ε, προδιαγραφές και να λάβουμε υπόψη παράλληλα και την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει ένα θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να συμμετέχουν οι πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η πρόταση κανονισμού για την διαφάνεια και την διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, Αποτίμησης Κινδύνων στην αλυσίδα τροφίμων αποτελεί ένα βασικό μας μέλημα για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των πολιτών και για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε τους κινδύνους. Η ε, βάση των αποφάσεών μας αφορά την ΕΦΣΑ, Θεωρώ ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός λοιπόν ε, Ασφάλειας Τροφίμων μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε υψηλά πρότυπα και πραγματογνωμοσύνη με βάση τις επιστημονικές μελέτες, μελέτες που έχουν ήδη διενεργηθεί και με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας διασφαλίζει την βελτίωση του συστήματος, το οποίο θα γίνει πιο εύρωστο και έμπιστο για την ασφάλεια τροφίμων. Θα θέλαμε να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτόν τον τομέα και έχω ε, αναλύσει τις ε, τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό τον τομέα. Πιστεύω λοιπόν ότι και το Συμβούλιο συμμερίζεται τους ίδιους στόχους σε σχέση με τα στοιχεία κλειδιά. Παρόλο που πολλές φορές υπάρχει διαφορετική διαφορετικό ε, πρίσμα αντιμετώπισης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πιλάρα Γιούσο για την διαθεσιμότητά της και γιατί ακριβώς συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για αυτό το ύψης της σημασίας ζήτημα. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, θα ήθελα να συνεργαστούμε στενά και να καταβάλουμε κοινή προσπάθεια για να φτάσουμε σε μια κοινή συμφωνία μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαχείριση με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν. Αυτή, αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λήθος για να φτάσουμε στην έγκριση του κανονισμού τον Μάρτιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η υγεία των ζώων επίσης είναι ύψιστο μέλημά μας γιατί συνεισφέρει και στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Η Ρουμανική Προεδρία θα αντιμετωπίσει τις μίζονες ασθένειες, ιδιαίτερα τις μολυσματικές ασθένειες που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Η Αφρικανική πανόλη των χείρων μας απασχολεί από το 2014 και ολοένα και διευρύνεται. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους και από οικονομικής άποψης. Η Ρουμανική Προεδρία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων και ε, θα γίνει μια διάσκεψη ειδικά για αυτή την ασθένεια στο Βουκουρέστι τους επόμενους μήνες. Σε τεχνικό επίπεδο, η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει συζητήσεις για μια συνεκτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την πρόληψη που να ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη εναρμονισμένα. Θα μας απασχολήσει η βιοασφάλεια για την πρόληψη των ασθενειών και την προστασία της υγείας των ζώων. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελε να θίξει η Προεδρία αφορά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής μέσα στα πλαίσια της ε, ενιαίας προσέγγισης της υγείας, One Health Approach. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να θέσουμε σε εφαρμογή τις σωστές πρακτικές μέσα στα πλαίσια της μικροβιακής αντοχής. Θα οργανωθεί στο Βουκουρέστι και μια υπουργική διάσκεψη. Η ευημερία των ζώων είναι ύψης της σημασίας επίσης για μας. Υπό αυτή την έννοια θα λάβουμε υπόψη τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για την ευημερία των ζώων και να ε, μειώσουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ στόχων και πρακτικής όπως δημοσιεύθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο στις 14 Νοεμβρίου 18. Οι εξαγωγές ζωντανών ζώων αποτελούν ένα βασικό έσοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρουμανική Προεδρία θα θέσει σε εφαρμογή τις καλύτερες πρακτικές για τις θαλάσσιες ιδιαίτερα μεταφορές. Οργανώνεται ένα σεμινάριο στο Βουκουρέστι τον Ιούνιο σε σχέση με τις εποπτικές αρχές και τις αρχές υγειονομικής επιθεώρησης. Μας ενδιαφέρει επίσης ο φυτοϊγειονομικός έλεγχος για την προστασία των φυτών και της ε, βιοπικιλότητας έτσι ώστε να μην, υπάρχουν, να μην υπάρχει επέκταση επιβλαβών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με τις καλλιέργειες, αλλά και τα μη καλλιεργήσιμα φυτά θα λάβουμε υπόψη την Διεθνή Σύμβαση Προστασίας των Φυτών μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού, της στρατηγικής μας 2020-30. Θεωρώ ότι ο τομέας της προστασίας των φυτών είναι ύψης της σημασίας γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές καθώς και την διεύρυνση και διάχυση των επιβλαβών οργανισμών. Γι' αυτό θα πρέπει να προλάβουμε την διάδοση αυτών των επιβλαβών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιβλαβών οργανισμών που πλήττει τα φυτά και φυσικά και τις ζωοτροφές. Η ξυλέλα φαστιντιόζα δημιουργεί μεγάλες ε, ζημίες στα φυτά ξενιστές στην Αμερική, Ασία και Ευρώπη. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι εάν αντιμετωπίσουμε το θέμα από πλευράς πρόληψης μακροχρόνια θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε αυτές τις ασθένειες. Οι δύο κανονισμοί, η Υγεία των Φυτών 2016-2031 και η επίσημη έλεγχη 2017 κάθετος 625 αποτελούν το ρυθμιστικό ευφυές πλαίσιο για μία πιο ασφαλή τροφή και ζωοτροφές μέσα στα πλαίσια και τη συνεργασία των εθνικών αρχών. Αυτή η πρωτοβουλία προωθήθηκε υπό βουλγαρική προεδρία και γι' αυτό θα προωθήσουμε διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μέρων έτσι ώστε να υπάρξει ο μέγιστος αντίκτυπος ε, ξεκινώντας από τον Δεκέμβριο του 2019 θα προωθήσουμε έναν εμβαθυμένο διάλογο όσον αφορά την υγεία των φυτών και την ευαισθητοποίηση των γεωργών και εξαγωγών εισαγωγών. Αυτή η δράση έχει πολύ μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε καλύτερα τον κίνδυνο αυτό των επιβλαβών οργανισμών καθώς και τις δράσεις και τα μέτρα για την συνολική υγεία των φυτών και για την ε, βιώσιμη παραγωγή και παραγωγικότητα. Το Διεθνές Έτος Υγείας των Φυτών 2020 αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να αρχίσουμε την εργασία μας ήδη από το 2019. Θα γίνει μια άτυπη συνεδρίαση των υπηρεσιών φυτοϊγιεινής τον Μάιο στην Κραϊόβα και θα δούμε ποιες θα είναι οι δραστηριότητες και τα μέτρα που προτείνουν τα, κρατά, τα κράτη με συγχωρείτε μέλη. Επίσης θα προωθηθεί μία διάσκεψη για την προστασία των φυτών και τις πολιτικές για τη δημιουργία μίας συγκεκριμένης δράσης πλαισίου για να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό για την παρουσίαση αυτή. Λοιπόν, ως είδηστε, συνάδελφοι, θα έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων, δύο λεπτά έκαστος οι συντονιστές και οι πρόσωποι των πολιτικών ομάδων και μετά θα απαντήσει ε, ο υπουργό αυτό τον πρώτο γύρο και θα ακολουθήσει δεύτερος με άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Πρώτος γύρος, η κυρία Γκροστέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για ε, να μας μιλήσετε. Περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Η Ρουμανική Προεδρία σας θα δει την ε, πρόοδο των εργασιών για την ε, μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ξέρετε ότι είμαστε πολύ προσιλωμένοι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των τροφίμων. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνουν ε, τους ε, αγρότες ε, για τους κινδύνους που διατρέχουν για να προστατεύουν το κλίμα και τα τρόφιμα. Και στην αιρεσιμότητα τη νέα δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία υποχώρηση στις απαιτήσει για το πρασίνισμα του προϋπολογισμού 2014-2020. Και αυτό δεν θα πρέπει να αφορά μόνο το κλίμα αλλά και τη βιοποικιλότητα και την καταπολέμηση της γενικής ρήπανσης. Ε, ποια είναι η άποψή σας για την ε, μετάβαση αυτή στην οικολογική εποχή της κοινή γεωρικής πολιτικής. Εργάστηκα επίσης πάρα πολύ ε, στον κανονισμό που αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα. Μας μιλήσατε για την αφρικανική πανόλη του χείρου και πώς βλέπετε αυτή την υπόθεση της εξάπλωσης της πανόλης του χείρου στην Ευρώπη και ποια είναι τα μέτρα που προτείνετε. Επίσης μας μιλήσατε για την αντοχή στα αντιβιωτικά, για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης, για την πάταξη αυτή είναι και προτεραιότητά σας. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες, ποιες δράσεις ακριβώς έχετε προβλέψει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπράνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και σας, Υπουργέ, που ήρθατε στην Επιτροπή μας σήμερα. Είναι δύσκολο να υπερβάλλει κανείς όταν μιλάει για την απειλή από την κλιματική αλλαγή. Εμείς τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, έχουμε πλήρη επίγνωση, τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα άμεσα και έμεσα. Και η πρώτη ερώτηση, παρόλο που ήρθε από άλλο πολιτικό κόμμα, αναφερόταν στην κλιματική αλλαγή, την οποία αφορά και δική μου ερώτηση. Η απειλή ε, βεβαίως έχει οξυνθεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε κάποιον στο Λευκό Οίκο, ε, που σημαίνει ε, ένα ε, γελοτοπιό, ο οποίος θεωρεί ότι εντάξει έπεσε και λίγο χιόνι και τι έγινε. Δεν υπάρχει καμιά κλιματική αλλαγή. Εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Και πολλοί κλάδοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, όπως ο ενεργειακός τομέας που έχει μειώσει τις εκπομπές. Υπάρχει όμως ένας κλάδος που μπορεί να έχει κάνει κάποιες ε, πρόοδους, αλλά υπολείπεται πολύ του επιθυμητού ε, και του εφικτού και αυτό είναι η γεωργία. Και ε, πραγματικά με κάθε εκταμίευση ε, ακούμε ότι θα υπάρχουν μειώσει στι εκπομπέ, γιατί είναι και τα χρήματα των φορολογουμένων που δεσμεύονται, αλλά δεν γίνονται αυτά με του ρυθμού και τι ταχύτητε που θα θέλαμε. Ανησυχώ λοιπόν Παρόλο που κάνετε μια εισαγωγή 18 λεπτών, δεν αναφερθήκατε ούτε στιγμή στην κλιματική αλλαγή και σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Ανησυχώ λοιπόν, ε, μήπως από πλευράς της Ρουμανικής Προεδρίας δεν είναι πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα αυτή η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Πήραμε τη μετάφραση ε, της άποψης της Γερουσίας τον Οκτώβριο του 2018 στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της ΚΑΠ και διαβάζοντάς τη δεν κατάλαβα ότι θεωρούν μεγάλη σημασία στην κλιματική αλλαγή ε, οι γερουσιαστές στην ε, Ρουμανία. Τα μέλη λοιπόν της Επιτροπής μας θέλουν να ε, μας επιβεβαιώσετε ότι ε, είναι ένα θέμα που σας απασχολεί αυτό και θα αξιοποιήσετε την Προεδρία σας για να βεβαιωθείτε ότι το επόμενο διάστημα, η προγραμματική περίοδος αυτή επταετής για την ΚΑΠ ε, στρέφεται και προς την κατεύθυνση αυτή. Τα Ηνωμένα Έθνη μας λένε ότι έχουμε μόνο 12 χρόνια για να αναστρέψουμε την κλιματική αλλαγή. Αν την επόμενη επταετία ε, στην ΚΑΠ την έχουμε ως περίοδο μεταβατική εντός εισαγωγικών, τι μας μένει, μια πενταετία για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Ε, δεν φτάνει αυτό, πρέπει να επιταχύνουμε. Και κάτι άλλο, ε, ενώ η κλιματική αλλαγή αποτελεί απειλή, αποτελεί και ευκαιρία μπορούν να δημιουργηθούν ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη βιοοικονομία που είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Δηλαδή εκτός από απειλή αποτελεί και ευκαιρία και μάλιστα ευκαιρία για πράσινες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεμές Μάκερ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και σας ευχαριστώ ειλικρινά για την εκτενή σας και εξαντλητική παρουσίαση. Δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Εδώ είμαι. Πρώτον, για το ρόλο της βιοτεχνολογίας στη γεωργία του μέλλοντος. Η βιοτεχνολογία είναι ένας τομέας σημαντικός για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι Φλαμανδός και η Φλάνδρα είναι μια περιφέρεια που έχει δείξει το δρόμο στην έρευνα συγκεκριμένα αυτή τη βιοτεχνολογική. Πιστεύω ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη φυτών που να αντιστέκονται σε κάποιες αρρώστιες ή και στην ξηρασία ή κάποια φυτά που να έχουν και περισσότερη απόδοση χωρίς να χρειάζονται περισσότερα λιπάσματα. Υπό την έννοια αυτή βλέπω και θεωρώ ότι η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι λίγο περίεργη, διότι απεφάνθη ότι οι νέες τεχνικές ε, εξευγενισμού, ε, το, η προσθήκη του γονιδιώματος genome editing θεωρείται ε, γενετική τροποποίηση. άρα αυτό έρχεται να καταπνίξει την ε, οποιαδήποτε καινοτομία και τεχνολογική πρόοδο στα σπάργανα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, η βιοτεχνολογία στην ε, γεωργική πολιτική που να είναι στραμμένη προς το μέλλον, έχει θέση, έχει νόημα και προγραμματίζεται στι τίποτα δράσεις. Ε, δεύτερη ερώτηση, πολύ σύντομα για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Αναφερθήκατε επιγραμματικά. Πέρσι η Επιτροπή μας εδώ περιβάλλοντος ενέκρινε μία γνωμοδότηση για την εκτέλεση του κανονισμού 1 του 2005, όπου βλέπουμε ότι η εφαρμογή του κανονισμού αυτού χωλαίνει, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Στο πρόγραμμα της Προεδρίας είδα κάποιες ε, αναφορές στην ε, προστασία της υγείας των ζώων στα σύνορα, αλλά δεν γίνεται λόγος ρητά για τις μεταφορές τους. Εσείς αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα στην εκτέλεση αυτού του κανονισμού και έχετε προγραμματίσει καμία δράση σχετικά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μιούλερ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, καταρχάς Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία ε, για την Προεδρία σας. Είναι δύσκολα τα πράγματα και τα θέματα που σας περιμένουν. Υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα που θέλουμε να τα έχουμε ολοκληρώσει πριν τις ευρωεκλογέ και αυτό χρειάζεται πηγόντως τη δική σας συνεργασία. Για ε, να προετοιμαστώ για τη σημερινή συνεδρίαση, διάβασα τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα θέματα. Ελπίζω όμως και τα θέματα της δικής μας Επιτροπής να μην ε, ξεχαστούν και να μην παραμεληθούν τους τελευταίους μήνες εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ασχολήθηκα εντατικά ε, με τη Γενική Νομοθεσία για το, τα τρόφιμα και την ΕΦΣΑ και στην Ειδική Επιτροπή ΠΕΣΤ που είχε συσταθεί για τα φυτοφάρμακα. Αναφερθήκατε λίγο στον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αλλά κατέληξα κι εγώ ότι στην ΕΦΣΑ ε, είναι πάρα πολύ αξιόλογα τα στελέχη εκεί και κάνουν και καταπληκτική δουλειά και θα πρέπει επιγόντως να φροντίσουμε να βελτιωθεί η χρηματοδότηση της ΕΦΣΑ, αλλά ε, να προχωρήσουμε και ε, με τους κανόνες για την επικοινωνία, ε, ενημέρωση των πολιτών όταν υπάρχουν κίνδυνοι, για να καταλάβουν οι πολίτες πόσο ασφαλή είναι τα δικά μας τρόφιμα και ποιες είναι οι διαδικασίες και οι μέθοδοι και πώς λειτουργούν για τον έλεγχο τους. Γνωρίζω ότι οι συζητήσει σε λεπτομέρεια δεν είναι πάντα εύκολε, αλλά το θέμα είναι τόσο σημαντικό, ε, ώστε να μην μπορεί να παραταθεί μέχρι μετά τις εκλογές. Ε, μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Και τέλος, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ασχολούμαι με αυτό ασχοληθήκαμε πάρα πολύ και εντατικά για την υγεία ε, πλαίσιο, για το πόσιμο είδο. Και περιμένουμε τώρα τη θέση του Συμβουλίου. Εχθέ είπε δύο λόγια ο συνάδελφο σα υπουργό Ιδάτων, αλλά σίγουρα τα γνωρίζετε κι εσείς και μπορείτε να μας ενημερώσετε γι' αυτά. Thank you very And Mr. How... Χόισλινγκ, ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Έχετε λίγο χρόνο, αλλά πολλά ε, θέματα που θέλετε να διεκπαιρεώσετε και έχουμε και τις ευρωεκλογέ. Στη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής πιστεύετε ότι πρόκειται να κινηθεί το παραμικρό πριν τις εκλογές. Έχω μεγάλες επιφυλάξεις, γιατί οι θέσεις των πολιτικών ομάδων απέχουν ακόμα πάρα πολύ από το Συμβούλιο και χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γίνει ο κανονισμός σωστός. Γιατί ε, σα το λέω και ειλικρινά, συμφωνώ και με τον Σνάιφο Μπράνεν, μου λείπουν εμένα κάποια πράγματα ακόμα. Η γεωργία για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του κλίματο έχει και αυτή να βάλει ε, το λιθαράκι τη. Δηλαδή, θα πρέπει και η γεωργία να έχει στόχου μείωση που δεν του βλέπω αυτή τη στιγμή. Και μετά η βιοπικιλότητα είναι κάτι που είναι ευθύνη και της γεωργίας και πρέπει να βρούμε λύσεις δεν μπορούμε να τα αναθέτουμε ε, σε κάποιες ε, περιοχές που είναι προστατευόμενες, δρυμή κτλ. Αλλά και στην ίδια τη γεωργία, στην κανονική γεωργία, να έχουμε λιγότερες παρεμβάσεις που απειλούν τη βιοπικιλότητα. Έχω και συγκεκριμένη ερώτηση. Ρώτησα και χθε τους συναδέλφους σας. Η Ρουμανία επικρίνεται σφοδρά, ε, διότι χάνονται δάση και σε εθνικά πάρκα και σε δρυμούς. Είπε ο συνάδελφός σας Υπουργό ε, Δασών ότι καλά δεν είναι και τόσο ε, φοβερά τα πράγματα. Ε, στην δασοκομεία υπάρχουν στόχοι όμως και τώρα είναι όλα εντάξει. Στη Ρουμανία βαίνουν καλώς. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη Γενική Νομοθεσία για τα τρόφιμα για να περάσει πριν τις εκλογές. Είναι κοινό ο στόχος αυτός ε, και το αποτέλεσμα της Επιτροπής ΠΕΣΤ για τα φυτοφάρμακα μπορούν πλέον να ε, τα αποτελέσματα μάλλον να ε, υιοθετηθούν και να εφαρμόζονται και να πούμε στις ευρωεκλογές ότι η διαφάνεια είναι βασικό αγαθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχουμε επιβάλει στην νομοθεσία για τα τρόφιμα. Ελπίζω να μας υποστηρίξετε εκεί και να προχωρήσουν και να έρθουν σε αίσιο πέραση οι διαπραγματεύσεις. Και ένα τελευταίο, συμφωνώ με τις προλαλήσαντες για τη μεταφορά ζών των ζώων. Είπατε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πώς θέλετε να τα λύσετε. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να διαφαίνεται καμία λύση. εκτός από το να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και διστακτικοί στο να μεταφέρουμε ζώντα ζώα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε ε, έναν μακρύ κατάλογο ερωτήσεων και μπορείτε τώρα να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά, τις περίμενα τις ερωτήσεις περίμενα γιατί ήρθα στο Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς ε, γι' αυτό το λόγο καθώς και στην αρμόδια επιτροπή αυτών των στόχων που αφορούν τους στόχους δηλαδή της ΚΑΠ. Μίλησα στην Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων γιατί μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων, για την τεχνολογική ασφάλεια και το σεβασμό του περιβάλλοντος για να ανταποκριθούμε στα ε, νόμιμα αιτήματα των καταναλωτών όταν μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν οι Ευρωπαίοι αγρότες και που χρησιμοποιούν ε, συγκεκριμένα μέσα υποστήριξης που προσφέρει η ΚΑΠ. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος των Ρουμάνων αγροτών που ευεργετήθηκαν πάρα πολύ από την ΚΑΠ και την οποία εκπονήσατε εσείς. Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε μια νέα ενιολογική βάση στην ΚΑΠ για την επταετία 21-27. Δηλαδή μια ΚΑΠ η οποία να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των αγροτών και στις προσδοκίες των πολιτών. Με βάση αυτή τη συλλογιστική και επειδή θέλουμε να είμαστε αρκετά πιστικοί και να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη ως προς το αναλυτικό μας σκεπτικό και την έμπρακτη δράση μας. Θα ήθελα να αρχίσουμε τις κλιματικές αλλαγές που σήμερα μας απασχολούν πάρα πολύ ως προς την ερμηνεία τους και τις επιπτώσεις τους. Οι κλιματικές αλλαγές δεν αποτελούν κάτι το άπιαστο, αλλά μία απτή πραγματικότητα. και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και από την ΚΑΠ για την επταετία 21-27. Θεωρώ ότι αυτή η ενιολογική βάση θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω και να βρεθούν τα υποστηρικτικά μέσα για να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση και ξέρουμε ότι θα έχει και επιπτώσεις για την επαύριο, χωρίς να ξέρουμε τις διαστάσεις επακριβώς των κλιματικών αλλαγών. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε έναν κοινό παρονομαστή με βάση τις επιπτώσεις και τη συνάφεια που αφορά μία οικολογική ζώνη ή ένα οικολογικό εύρος θα μπορούσα να πω, για να δώσουμε απάντηση στα θεμητά ερωτήματα των πολιτών. Πώς βλέπουμε δηλαδή αυτές τις αγροτικές δραστηριότητες που πλαισιώνονται από τα βασικά μελήματα των καταναλωτών και των καλλιεργητών. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους αγρότες, τους παραγωγούς, αλλά να κρατήσουμε τη βιοπικιλότητα με βάση την ε, καθημερινή ζήτηση και προσφορά και λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πρόσταγμα του να είναι κανείς παραγωγός τροφίμων, ε, τροφίμων που αποτελούν, που μάλλον παρέχουν προς προδιαγραφές ασφαλείας. Οι κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να τύχουν μιας ευφυούς αντιμετώπισης και συνέργειας με βάση επιστημονικά στοιχεία για να παρακολουθήσουμε τις βιοτεχνολογικές αλλαγές μέσα στα πλαίσια ε, μιας γενικότερης αρμονίας ανθρώπου φύσης και φυσικά και όλων των προαπαιτούμενων που προβάλλει ο πολίτης και ο καταναλωτής. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε αυτή την ε, υποστήριξη μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ και των ε, μελημάτων του πολίτη. για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, τις παρούσες προκλήσεις. Σε σχέση με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τις ε, μεταλλάξεις και εδώ θα πρέπει να ερμηνεύσουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κάτι το οποίο αφορά μέσα τους αγρότες και τους παραγωγούς γενικότερα και γι' αυτό χρειαζόμαστε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για να αντιμετωπίσουμε τις ε, τις φυσικές μεταλάξεις και τις τεχνητές. Να γίνει δηλαδή αυτή η διαφοροποίηση. Χρειάζονται διασαφηνίσεις και στον ε, τομέα των βελτιώσεων, διότι οι κλιματικές αλλαγές οδηγούν και σε μία νέα τεχνολογική προσέγγιση. Έτσι δίνουμε μία νέα όθηση στην ΚΑΠ με συγκεκριμένες προσαρμογές και με βάση πρωτεϊνούχα ε, φυτά τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν και στην μείωση των ρήπων. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε ενεργά για να υποστηρίξουμε την έρευνα και τη διαδικασία βελτίωσης έτσι ώστε με βάση αυτή τη διαδικασία να έχουμε ε, μία αυξημένη αντίσταση και αντιμετώπιση για παράδειγμα της ξηρασίας και επίσης να αντιμετωπίσουμε τους επιβλαβείς οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις επιπτώσεις ορισμένων σοβαρών ασθενειών, όπως η ξυλέλα φαστιντιόζα. Επίσης, φυσικά ε, μπορεί να υπάρξει επίπτωση και επί της παραγωγής από 30 έως 80% με βάση την δράση αυτών των επιβλαβών οργανισμών. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και αποφάσεις και να υπάρχει μία εξισορροπημένη προσέγγιση των αγροτών και παραγωγών για την ασφάλεια τροφίμων και τον σεβασμό της φύσης και της βιοπικιλότητας. Με άλλα λόγια, αυτά τα μέτρα συνέργειας είναι ύψης της σημασίας και μας απασχολούν και σε νομικό επίπεδο. τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να προωθήσουν αυτά τα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε θέματα που άπτονται της γεωργίας αλλά και όχι μόνο. Συμφωνούμε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και παρακολουθούμε το θέμα εκ του σύνεγγης σε σχέση με τις μελλοντικές μας πολιτικές στο τομέα της ε, βιοτεχνολογίας. Σε σχέση τώρα με την ε, ε, μικροβιακή αντοχή στα αντιβιωτικά, η Ρουμανική Προεδρία θα συνεισφέρει στην καταπολέμηση αυτής της μάστιγας και γι' αυτό το λόγο η Ρουμανική Προεδρία θα οργανώσει μία ε, διάσκεψη για την καταπολέμηση της ε, μικροβιακής αντοχής στα αντιβιωτικά και θα δούμε ποια θα είναι τα συμπεράσματα αυτής της ε, διάσκεψης. Εδώ πολύ σωστά αναφέρθηκαν πολλές ανησυχίες Μιλήσαμε για την ε, συνείδηση, επαγγελματική συνείδηση των επιστημόνων, στη συνείδηση των αγροτών και στην αντιμετώπιση της αφρικανικής πανόλης των χείρων. Η Ρουμανία γνώρισε αυτή την ασθένεια. Εδώ και πέντε χρόνια, μάλλον κατά διάρκεια πέντε ετών, 12-17, μεταξύ 2012 και 2017, κλείσαμε τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και μιλάμε για μία απόσταση για ένα μήκος 1.400 χιλιόμετρων. Ε, αυτό το μικρόβιο μπήκε από μία ε, ζώνη, από μία περιφέρεια που γνωρίζετε πολύ καλά και εμείς ε, καταφέραμε... Delta Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βιοπικιλότητας και της αντιμετώπισης της πανόλους γιατί ακριβώς ε, κλείσαμε τα σύνορα και γι' αυτό περιορίσαμε την εμβέλεια του ιού παρόλο που μπήκε, διείσδησε στα σύνορά μας, εν πάση περιπτώσει τον αντιμετωπίσαμε με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιμετωπίσαμε το θέμα της διάδοσης του σε αρκετές περιφέρειες της Ρουμανίας. Περιορίσαμε λοιπόν τον ιό, τον αντιμετωπίσαμε με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων και με την αρρωγή της Επιτροπής. Με ειδικού από όλο τον κόσμο που σήμερα βάσει της πείρας τους μπορούν να μας δώσουν τα κατάλληλα ε, χέγγια και στοιχεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας θα γίνει μια διάσκεψη στο Βουκουρέστι για αυτό το θέμα. Άρα προσδίδουμε μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας και επενδύσει στον τομέα της έρευνας έτσι ώστε στο εγγύς ε, μέλλον να βρούμε μία απάντηση για να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι υπάρχει κοινό ενδιαφέρον και από εσάς και από εμάς, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος μας εχθρός. Εμείς λοιπόν, μέσα στα πλαίσια της Προεδρίας και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους ειδικούς εμπειρογνώμονες και ούτω καθεξής, θα αντιμετωπίσουμε και θα περιορίσουμε παρόμοιες ασθένειες. Θα υπάρξει και ένας θεσμικός διάλογος για θέσουμε σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα και τις προτεραιότητες που σας παρουσίασα σήμερα. Οι κλιματικές αλλαγές μας απασχολούν εκ του σύνεγγυς και φυσικά γνωρίζουμε ότι αποτελούν μία απτή πραγματικότητα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους μας. Παράλληλα, θα ήθελα να σταθώ στην υποστήριξη των αγροτών με βάση ορισμένες ε, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για να παρακολουθήσουμε την καθημερινή τους εργασία και να τους ε, ε, δώσουμε τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσουν τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες που πλήττουν την παραγωγή και που φυσικά τους υποχρεώνουν να αναλάβουν το κόστος αυτών των ασθενειών πολλές φορές και των αρνητικών επιπτώσεων. Πολλοί έθεσαν ερωτήματα σε σχέση με τη δυνατότητα ανταπόκρισης στα ζητήματα που μας αντιμετωπίζουν, που, μας, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, συγγνώμη, και τώρα και στο μέλλον, καθώς και τις συγκεκριμένες δράσεις με άμεση συνεργασία και συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Κατά την προσεχή περίοδο θα έχετε τη δική μας ανταπόκριση και άμεσες απαντήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες. Και ελπίζουμε να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών και αναγκών μέσα στα πλαίσια και της άμεσης συνεργασίας με τις άλλες επιτροπές που ασχολούνται με παρόμοια ζητήματα, δηλαδή ε, και την Επιτροπή Άγκρη, όπου αύριο θα παρουσιάσω τις προτεραιότητες μας. γιατί φυσικά το Συμβούλιο γνωρίζει το εύρος των ζητημάτων και ελπίζουμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις γνωρίζοντας τις ανάγκες των αγροτών και των ε, παραγωγών. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Παρακαλώ, ένα λεπτό ο καθένας. First one ε, is Madame Κυρία πρώτη. Ευχαριστώ. καλώ ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Κάνατε μια αρκετά μακροσκελή παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας, αλλά μια και μιλάτε για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, θέση την οποία λάβατε για την ε, καινούργια ΚΑΠ σε ό,τι αφορά την ε, οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητά της και πιο συγκεκριμένα για την ε, δυνατότητα το περιβάλλον να γίνει ευκαιρία για τον αγροτικό κόσμο και να μην έρχεται συνεχώς σε αντίθεση η γεωργία με το περιβάλλον, να μην συγκρούονται. Ε, ένα από αυτά τα θετικά θέματα είναι το ε, πλάνο για τις πρωτεΐνες θα μπορούσαμε να ε, καλλιεργήσουμε πρωτεϊνούχα φυτά ε, για, να, για ζωοτροφή ε, και για καύσιμο, έτσι ώστε να απο... έτσι ώστε να αποφύγουμε να εξαρτώμαστε από εισαγωγές. Το είπε και ο ε, Θέλω να επιμείνω. Θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές ε, έναντι της ε, χρήσης ε, φυτοφαρμάκων με τις νέες βιο... τεχνικές της βιοτεχνολογίας. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω. Κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το επόμενο εξάμεινο και έχετε να αντιμετωπίσετε μεγάλες προκλήσεις για την ΚΑΠ. Το νέο πακέτο μετά το 2021 αποτελεί μια νέα πρόκληση για τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε σχέση με την οικολογική διάσταση greening της ΚΑΠ. Μπορείτε να μας πείτε ότι το Συμβούλιο θα προωθήσει βιώσιμες πρακτικές. Δεν θα γίνει η επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Μπορείτε να μας το εξασφαλίσετε αυτό, να μας το εγγυηθείτε. Θα υπάρξει πραγματικά το πρασίνισμα, το επωνομαζόμενο της ΚΑΠ όπως επιθυμούμε όλοι. Ο κύριος Σκάνου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω και εγώ, να σας ευχηθώ και εγώ κάθε επιτυχία. Μιλήσατε για 20 λεπτά, 20 λεπτά και δεν μας απαντήσατε άμεσα. Η κυρία Γκροστέτ σας μίλησε για την οικολογική γεωργία και εσείς δεν είπατε τίποτα απολύτως τίποτα. Θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας. Το θέμα το έθεσε κυρίως η κυρία Γκροστέτ. Υπάρχει και το πρόγραμμα ε, LIFE, το οποίο διαθέτει πάρα πολλά χρήματα και εντάσσεται στη Natura 2000. Ε, η Ρουμανία έχει μία επιφάνεια που το 1 τρίτον αφορά δασοκομικές ε, δάση μάλλον, δασολογικές, δασολογικές εκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο έδαφος ε, σχετίζεται με την αγροτική οικονομία. Μπορείτε να μας πείτε ποιες θα είναι οι αντισταθμίσεις που θα δοθούν στους ε, γεωργούς Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση των αντισταθμίσεων και ποια είναι η απάντησή σας. Ευχαριστώ κυρία Σχράιερ Πύρικ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του. Ε, θέλω να μιλήσω για την αντοχή στα ε, αντιβιωτικά. Εγώ προετοιμάζω τώρα μία ε, διάσκεψη και εσείς εσείς έχετε καλέσει το Κοινοβούλιο, τους Υπουργούς, ε, ήταν και η κυρία Γκροστέτ που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Ωραία, έγινε αυτή η διάσκεψη και τι συνέχεια θα δώσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη Γεωργία φυσικά και για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, για την Πανόλη του Χείρου θέλω να ρωτήσω. Τι γίνεται με τις ιατρικές εξελίξεις και τις φαρμαλογικές. Δεν μπορούμε να το λύσουμε το θέμα αυτό διαμαγείας. Και να πω και κάτι άλλο για το λύκο. Συχνά έχουμε προβλήματα με τους λύκους στην Ευρώπη και θα πρέπει να διαχειριστούμε. Εμείς ε, ξέρουμε και εσείς έρχεται από, ε, από μια χώρα ε, που έχει πολλούς λύκους και υπάρχει πρόβλημα για τα πρόβατα και για διάφορα πτηνά και τα λοιπά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Ο συνάδελφος Ντόρφμαν έχει καταθέσει σχετικό ψήφισμα για το λύκο. Ευχαριστώ κύριο Σπαρνιό. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Όπως αναφέρθηκε και όπως είπε η κυρία Τελαέ, ε, η καινούρια ΚΑΠ ε, θα, θα εξεταστεί από το καινούριο κοινοβούλιο και σίγουρα θα πρέπει να περιλαμβάνει και την... Ε, τα τρόφιμα και την ασφάλεια των τροφίμων. Γι' αυτό το θέμα, στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας 17 και 18 Δεκεμβρίου 2018, η Γαλλία πρότεινε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ομάδας έρευνας για την ε, διαρεύνηση και για την καταπολέμηση των τροφιμικών ε, επιγόντων περιστατικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ρουμανική Προεδρία σκοπεύει να προωθήσει αυτή την πρόταση της ε, δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Μονάδας Έρευνας και Ελέγχου τα επόμενα, τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, η μικροβιακή αντίσταση, αντοχή στα α, ε, αντιβιωτικά αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν τα εθνικά συστήματα υγείας αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα. Και αυτό αφορά άμεσα τη γεωργία γιατί δυστυχώς ε, γίνεται άλογη χρήση των ε, αντιβιωτικών για λόγους προφύλαξης, κάτι το οποίο ακριβώς οδηγεί σε αυτή την μικροβιακή αντοχή. Πιστεύω λοιπόν ότι οι Υπουργοί Υγείας θα πρέπει να προσκληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Γκροστέτ έχει προωθήσει μια μεγάλη εκστρατεία ως προς αυτό το θέμα που αποτελεί προστιθέμενη αξία. Τώρα, σε σχέση με την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, πώς βλέπετε να γίνει μία ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Γιατί δυστυχώς ε, στη Ρουμανία υπάρχουν ολοένα και περισσότερα κρούσματα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μπράνεν έχει το λόγο. Μια σύντομη ερώτηση μόνο ε, μίλησαμε για τα μεγάλα σαρκοβόρα και τώρα μιλάμε και για τους λύκους. Ε, έχει γίνει μια μελέτη από την Σλοβακία που δείχνει ότι όπου υπάρχουν λύκοι δεν υπάρχει ε, ε πανόλη χείρων. Οπότε προφανώς υπάρχουν επιχειρήματα κατά των λύκων, αλλά υπάρχουν επιχειρήματα και υπέρ των λύκων. Κύριε Υπουργέ, έχετε πάλι το λόγο για ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων. Ναι, είναι απόλυτα φυσικό και απόλυτα αναγκαίο θα μπορούσα να πω. Σε σχέση με τα πρωτεϊνούχα φυτά, ε, αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της Ουρμανικής Προεδρίας. Έχουμε συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα και φυσικά και την θέση των αγορωτών. Τη στιγμή που γίνεται χρήση φυτοφαρμάκων, ευρεία χρήση, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να ε, συρρυκνωθεί, να περιοριστεί αυτή η χρήση μελλοντικά, για να δούμε ποια θα είναι και η ε, ανταπόκριση των αγροτών. Τι βάζουμε όμως στη θέση αυτών των ε, φυτοφαρμάκων. Θα πρέπει οι αγρότες να γνωρίζουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να υπάρχουν αντισταθμίσματα. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη χρήση αυτών των ε, φυτών θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό, αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Η Ευρώπη καταναλώνει όλο ένα και περισσότερο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σόγια η οποία εισάγεται από αλλού. Και δυστυχώς αυτό αφορά τους γενετικώς ε, τροποποιημένους οργανισμούς. Γι' αυτό στις 28 του μήνα θα ασχοληθούμε ακριβώς με αυτά τα πρωτεϊνούχα φυτά για να μπορέσουμε να σφυριλατήσουμε μία νέα πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση για να υποστηρίξουμε την ΚΑΠ και για να αυξήσουμε αυτό το φάσμα των πρωτεϊνούχων φυτών. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες έτσι ώστε να ε, περιορίσουν την χρήση των παρασιτοκτόνων και των φυτοφαρμάκων. Και αυτό αφορά και πολλές καλλιέργειες όπου υπάρχει μικροβιακή αντίσταση. Και για να έχουμε τα κατάλληλα τρόφιμα, τη σωστή παραγωγή και την ασφαλή παραγωγή τροφίμων με την υποστήριξη βεβαίως των αγροτών και για να υπάρχει και εξασφαλισμένη τροφή ενώ παράλληλα θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να εισαγάγουμε αυτά τα φύτα, αυτή την, δηλαδή την οικολογική προσέγγιση γιατί το γονιδίωμα των φυτών είναι τέτοιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει φυσικούς παράγοντες χωρίς ε, χημικά, χωρίς χημικές ουσίες. Για να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις αυτές σε σχέση με το οικολογικό μας μέλημα. Αυτό αποτελεί άμεση ανησυχία όλων και της Ρουμανικής Προεδρίας. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες πρωτεϊνούχες ουσίες για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι επιβλαβείς παράγοντες. Θα δοθούν λοιπόν απαντήσεις με βάση τις αρμοδιότητες που διαθέτουμε στο Συμβούλιο Υπουργών και τα κράτη-μέλη θα συνδράμουν για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά θα ήθελα να πω ότι και ο επιστημονικός κόσμος ε, θα συνδράμει έτσι ώστε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό τον τομέα με συγκεκριμένα μέτρα Και αυτό αφορά και τη Natura 2000, έχοντας πρόσβαση στους ε, κατάλληλους πόρους, όπως είπατε και εσείς. Da? Unitate de forță. Ισχύσεν τη ενώση. Έτσι θα πρέπει να δράσουμε. Θα λάβουμε υπόψη την πρόταση που προέρχεται από τη Γαλλία. Θα συναντηθώ άμεσα με τους συναδέλφους, αλλά παράλληλα εκτιμώ το γεγονός ότι η απόφαση αυτή θα μπορέσει να ληφθεί παράλληλα με τα άλλα κράτη, από κοινού με τα άλλα κράτη, γιατί όλοι συμπαρασυρώμαστε προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στα πλαίσια κοινού ενδιαφέροντος και συμφερόντων. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πολύ σωστό επιχειρησιακό πλαίσιο. Αλλά καταρχήν θα καλέσουμε στη Ρουμανία στις διασκέψεις αυτές και τους ευρωβουλευτές από τις αρμόδιες επιτροπές. Γιατί κατανοούμε απόλυτα αυτή την ανάγκη συνδρομής από τους καθήλυν αρμόδιους και φυσικά οι λύσεις βρίσκονται με τη συνδρομή όλων, μαζί με όλους και διαμέσου όλων. Θα σας στείλουμε λοιπόν προσκλήσεις για τις αντίστοιχες ε, διασκέψεις και σεμινάρια. και θα ήθελα να σας καλέσω να έρθετε στη Ρουμανία σε αυτές τις συναντήσεις για να γίνει μία ευρεία συζήτηση για τα θέματα τα οποία φίξατε και εσείς σήμερα. Και φυσικά θα καλέσουμε και επιστήμονες και εμπειρογνώμονες για να γίνει μία ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για να θέσουμε σε εφαρμογή τα σχέδιά μας και για να επιτύχουμε για αυτόν ακριβώς το λόγο. de Καρνιβόρη Σε σχέση με τα μεγάλα σαρκοβόρα, των πληθυσμό τους. Αυτό αποτελεί θεμητό ερώτημα και ανησυχία όλων των κρατών ε, μελών και γι' αυτό η Ρουμανική Προεδρία θα προσπαθήσει, θα προσπαθήσει να ε, ανταποκριθεί, με, θα συναντηθούμε στα πλαίσια της ΚΟΠΑ και της ε, ΚΟΤΖΕΚΑ για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Πρόκειται για κοινή ανησυχία για να δούμε ποια οδό θα πρέπει να ακολουθήσουμε χωρίς βεβαίως να χαλάσουμε την ισορροπία της ε, βιοπικιλότητας έμπρακτα. Αλλά να λάβουμε υπόψη και το θεμητό μέλημα των αγροτών και των εκτροφέων. Γιατί υπάρχουν, ε, δυστυχώς ε, προκύπτουν μεγάλες ζημίες και μεγάλες ανησυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία κατά την Ρουμανική Προεδρία για να αντιμετωπίσετε τα θέματα που μας απασχολούν όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνεται εδώ η πρωινή συνεδρία. Σε ραντεβού το απόγευμα με την Υπουργό Υγείας στις 2.30. Ευχαριστώ πολύ.